colleagues, uh, we're running Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω μια μικρή καθυστέρηση, γι' αυτό δεν θα ήθελα να χρονοτριβούμε άλλο. Παρακαλώ καθίστε και θα ήθελα στο επόμενο λεπτό να αρχίσουμε. Right, could we now begin? κύριε, την έναρξη της συνεδρίασής μας. Καλημέρα σας και ζητώ συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση, γιατί οι επιτροπές ε, Λίμπε και ΑΦΕΤ συνεδρίασαν από κοινού και δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε εγκαίρως την κοινή μας αυτή συνεδρίαση. Περνάμε τώρα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά την κυρία Γκαβριέλα Κουέβας Βαρών, και να την ευχαριστήσω που ήρθε στη συνεδρία. Σε λίγο θα συζητήσω μαζί της ένα θέμα. Επίσης να καλωσορίσω τον πρέσβη του Μεξικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συνοδεύει την κυρία Κουέβας Μπαρόν. Θα ήθελα να προσθέσουμε στην ημερήσια διάταξη στο σημείο 16 μία ενημέρωση για τις βουλευτικές εκλογές που έγιναν στο Κωσυφοπαίδιο στις 6 Οκτωβρίου. Συμφωνείτε? Ωραία. Οπότε η μερίσια διάταξη εγκρίνεται αφού δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Σημείο 3. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Τρει ανακοινώσει έχω. Η πρώτη αφορά το γεγονό ότι δεν έχει οριστεί ακόμη επίτροπο για την διεύρυνση και την πολιτική γειτονία, οπότε δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η ημερομηνία τη ακρόση μαζί του. Πολλοί συνάδελφοι ενδιαφέρονται για το πότε θα γίνει η ακρόαση, οπότε έχουμε στοιχεία, θα σας ενημερώσουμε. Και εγώ είμαι πολύ περίεργος για το πότε θα γίνει τελικά αυτή η ακρόαση. Δεύτερον, η προθεσμία για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με το Βιετνάμ και την Συμφωνία Προστασίας των Επενδυτών άλλαξε από τις 13 Νοεμβρίου το μεσημέρι ε, ε ε, ε, μετατοπίστηκε στι 13 Νοεμβρίου μάλλον, γιατί η 11η Νοεμβρίου είναι αργία, οπότε δεν θα μπορέσουν πολλοί να έρθουν εγκαίρως και να καταθέσουν τροπολογίε στι χρωμοδοτήσεις, όπω σας ανέφερα προηγουμένω εμπρόθεσμα. Γι' αυτό παρατείνεται κατά δύο ημέρε. Ο κύριο Κιουτσουκ ε, από την ομάδα Ρινιού, ζήτησε το λόγο για την ασφαλή επιστροφή του κυρίου Ρένση και άλλων μελών της αντιπολίτευσης από την Καμπότζη ε, ζήτησα το λόγο για την πολιτική κατάσταση στην Καμπότζη και κυρίως του Σαμ Ρέμζη, ε, από τους αρχηγούς αντιπολίτευσης και ε, ως ομάδα ετοιμάσαμε μία σύντομη δήλωση, τη στείλαμε στην ΑΕΔ. Ε, σας την έχουμε στείλει και ηλεκτρονικά και ζητούμε να μας υποστηρίξετε για να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στην Καμπότζη. Ευχαριστούμε κύριε Κιουτσούκ για την ενημέρωση. Έχετε άλλα σχόλια? Όχι, οπότε περνάμε στο σημείο 4, την έγκριση των πρακτικών των τελευταίων μας συνεδριάσεων της 10ης Ιουλίου, 24ης Ιουλίου, Δευτέρας και 3 η Σεπτεμβρίου και 8ης Οκτωβρίου. Έχουμε μοιράσει τα πρακτικά, οπότε αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, προτείνω να τα εγκρίνουμε όσα έχουν. Και περνάμε τώρα στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης και να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο Βαστσικόφσκι για να προεδρεύσει σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων με την Πρόεδρο της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης. Ευχαριστώ, Ντέιβιτ, και καλημέρα σας. Ε, με ιδιαίτερη περηφανία και τιμή καλωσορίζω την κυρία Καμπριέλα Κόβας Μπαρόν, την Πρόεδρο της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης. Η κυρία Κόβας Μπαρόν είναι μεξικανή βουλευτής και εξελέγει στην Προεδρία της ε, Διακοινοβουλευτικής Ένωσης με τριετή θητεία το 2017. Προεδρεύεται, κυρία μου, ε, μια οργάνωση 130 ετών, στην οποία συμμετέχουν 179 εθνικά κοινοβούλια και το, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καμαρώνει γιατί είναι συνδεδεμένο μέλος και συνεργάζεται μαζί σας ε, για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνουν και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα. Ε, κυρία Κόβας Μπαρόν, τα κοινοβούλια είναι η ραχοκοκαλιά της δημοκρατίας και το έργο του υπερβαίνει ε, το νομοθετικό, εποπτικό και δημοσιονομικό τομέα. Και στι εξωτερικέ υποθέσει, η κοινοβουλευτική δημοκρατία προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο νομιμοποίηση στη διακοινοβουλευτική συνεργασία. Ο ρόλο των, των βουλευτών είναι να προωθήσουν το διάλογο, την ειρήνη και το κράτος δικαίου σε εθνικό αλλά και υπερεθνικό επίπεδο. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, διαβιούμε σε δύσκολους καιρούς όπου η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πολυμέρεια και η ειρήνη δοκιμάζονται. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης ε, που βοηθά τους, τους κοινοβουλευτικούς να ενισχύσουν τη δημοκρατία είναι σημαντικότερο από ποτέ. Από αυτή την άποψη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να διευρύνει τις δραστηριότητες του στήριξη δημοκρατίας, όπως είναι η παρατήρηση εκλογών, η δημιουργία κοινοβουλευτικών ικανοτήτων και οι πρωτοβουλίες διαμεσολάβησης. Και μάλιστα ε, χαιρόμαστε που είστε εδώ μετά την 141η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής ε, Ένωσης που έγινε στη Σερβία στα μέσα Οκτωβρίου 2019 και εστιάστηκε στην ενίσχυση του διεθνούς δικαίου. Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο κυρία Πρόεδρε για περίπου 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε Μακάλιστερ, ευχαριστώ κύριε Βασικόφσκι για την ευκαιρία αυτή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Θα μιλήσω στα ισπανικά, στη μητρική μου γλώσσα. Οι επίσημες γλώσσες μας είναι αγγλικά και γαλλικά, αλλά αισθάνομαι πολύ πιο άνετα να μιλήσω στα ισπανικά. Η Κοινοβουλευτική Ένωση, όπως ε, λέγατε και εσείς, εκπροσωπεί 179 χώρες και κοινοβούλια. Υπό την προώθηση της δημοκρατίας, την πράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουμε ψηφίσματα, διακηρύξεις και συζητήσεις. Στην πραγματικότητα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα όλοι οι κοινοβουλευτικοί σημαντικές προκλήσεις, ιδιαίτερα εκείνοι που δουλεύουμε στα πλαίσια της πολυμέρειας. Έχουμε μια συνεργασία λοιπόν και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε την διακοινοβουλευτική διάσκεψη για θέματα παγκοσμίου εμπορίου. Εκπροσωπείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις ολομελιές μας. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε διάσκεψη στην Ιαπωνία με το P20 των προέδρων δηλαδή των κοινοβουλίων των 20 πιο ανεπτυγμένων χωρών στην, στον κόσμο. Και πολύ χαίρομαι που μπορούμε να συζητούμε και να συνεργαζόμαστε, μοιραζόμαστε την πρόθεση του να δώσουμε μια νέα προώθηση και να υπερασπίσουμε την πολυμέρεια, γιατί βλέπουμε σήμερα περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν ότι δεν μπορούμε να παραχωρούμε περιθώριο έναντι της προάσπισης των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σχετικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των νέων, όλα αυτά θα πρέπει να μετατραπούν σε πραγματικότητα. Και μπορούμε να πούμε ότι πράγματι τα κοινοβούλια είναι η καρδιά της δημοκρατίας, καρδιά όμως που σήμερα δεν εκπροσωπεί τους πολίτες όπως τα θέλαμε. Άνω του μισού του παγκόσμιου πληθυσμού είναι γυναίκες, αλλά μόνο το 24% των κοινοβουλευτικών εδρών κατέχονται από γυναίκες. Πάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού έχει 30 έτη ηλικία, αλλά μόνο περί το 1, το 2,2% του, των παγκοσμίων εδρών αντιστοιχεί σε αυτήν την ηλικία. Επίσης υπάρχουν κοινοβούλια που δεν επιτρέπουν καν να είναι κανείς υποψήφιος όταν είναι νεαρότερος των 30 ετών. Εάν θέλουμε λοιπόν τα κοινοβούλια πραγματικά να αποτυπώνουν την κοινωνία και βλέπουμε διαδηλώσεις και ανησυχία και δυσαρέσκεια στον κόσμο, πρέπει να αποτυπώνουμε την κοινή γνώμη. Ε, οι, περισσότεροι, οι περισσότερες από τις χώρες που εκπροσωπούμε έχουν ήδη μια δημοκρατική παράδοση. Αντιλαμβανόμαστε όμως τι είναι να μάχεται κανείς για τη δημοκρατία. Οι νεότερες γενιές ίσως το αντιλαμβάνονται πιο δύσκολα. Είναι ε, δύσκολο να φανταστεί κανείς τι συνέβη κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Σήμερα έχουμε την τεχνολογία με την αμεσότητα που μας επιτρέπει να έχουμε ενημέρωση πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά και με τις απειλές που δεχόμαστε από τον λαϊκισμό τις προκλήσεις κατά της δημοκρατίας, τον εθνικισμό. Έχουμε την αφήγηση, την σύγκρουση αν θέλετε, την διαλογική μεταξύ του, πολυ... της πολυμέρειας και της μονομέρειας και πρέπει να βρούμε λύσεις και συνενετικές απόψεις. Πρέπει να βρούμε ισορροπίες μεταξύ του προστατευτισμού και της ελεύθερης οικονομίας, των ελεύθερων συναλλαγών. Την ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και της ασφάλειας. της ανοχής και της ξενοφοβίας, της ανοιχτή κοινωνίας και της κλειστής κοινωνίας. Ε, είναι προβλήματα που θεωρούσαμε ότι είχαμε αφήσει πίσω μας μετά τους πολέμους του 20ου αιώνα. Αλλά εδώ βρισκόμαστε. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι πρέπει καταρχάς να αναλύσουμε απολύτως ειλικρινά το τι συμβαίνει σήμερα στον πλανήτη μας και που ενδεχομένως δεν εκπροσωπείται σήμερα η πλειοψηφική άποψη των πολιτών. Αν θέλει κανείς σήμερα να δει ένα έργο, να αγοράσει ένα προϊόν, ένα αγαθό, αρκεί πολύ συχνά ένα τηλέφωνο ή μια πιστοτική κάρτα. Αυτή η αμεσότητα όμως δεν μεταφεράζεται στις ε, πολιτικές, στις δημόσιες πολιτικές, οι προσδοκίες μεγάλου μέρους του πολιτισμού για άμεση κάλυψη των αναγκών του δεν υλοποιείται μέσω της πολιτικής ζωής, του πολιτικού βίου. Και αυτή η αναντιστοιχία οδηγεί σε καχυποψία τους πολίτες. Πολλοί νέοι δεν κατανοούν γιατί δεν μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά μας. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε πιο αντιπροσωπευτικοί τη κοινωνία, τη κοινή γνώμη όταν λαμβάνουμε αποφάσει. Και έχω την εντύπωση ότι σήμερα, στον 21ο αιώνα και με 30 χρόνια ιστορία στην διακοινοβουλευτική και 130 με συγχωρείτε χρόνια ιστορία στην Διακοινωνιστική Ένωση, πρέπει να βρούμε νέα πρότυπα διακυβέρνησης που να μπορούν να δίνουν λύσεις, να δίνουν απαντήσεις, να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του κόσμου που εκπροσωπούμε. Μπορούμε να αναρωτηθούμε γιατί είναι τόσο της μόδας σήμερα να ακούμε επικρίσεις κατά του συστήματος πολυμέρειας, γιατί βλέπουμε διαδηλώσεις δυσαρέσκεια. Πρέπει να βρούμε νέους χώρους συμπερίληψη συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης απόφασης. Πρέπει να έχουμε τον άνθρωπο στο κέντρο της προσπάθειάς μας. Τον πραγματικό άνθρωπο, τον απτό άνθρωπο. Όχι απλώς να ασχολούμαστε με εκστρατείες ε, εκλογικές ή στατιστικά δεδομένα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ένωσης του χρόνου τον Αύγουστο θα έχουμε την πέμπτο, το πέμπτο συνέδριο των Προέδρων των Κοινοβουλίων. Αυτό συμβαίνει μόνο κάθε πέντε χρόνια. Και είναι βήματα όπως αυτό στα οποία μπορούμε πραγματικά να αναπτύξουμε ποιο είναι το μέλος του κοινοβουλευτικού συστήματος, του κοινοβουλίου ώστε να είναι πιο ζωντανό, πιο κοντινό στον κόσμο και να ξαναδώσει εμπιστοσύνη στους πολίτες. Εγώ θα έκλεινα εδώ την εισαγωγή μου ώστε να έχουμε και χρόνο για ερωταπαντήσεις. Έχουμε πολλές σκέψεις, πολλές ιδέες για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε η Διακοινοβουλευτική Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι κοινή η πρόθεσή μας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία. Έχουμε κοινέ απόψεις και, έχουν, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως μπορεί να μας βοηθήσει σε θέματα παρακολούθησης εκλογών, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε σε θέματα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων γυναικών, της ισότητας των φύλων και του θεματολογίου ανάπτυξης του 2030. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μαζί σας και ελπίζω να συναντιόμαστε και πιο συχνά στο μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you very much, Madam President. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την εισήγησή σας προχωρήσουμε στη συζήτηση. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συντονιστές. Ε, ο πρώτος ε, στον ε, κατάλογο των ομιλητών είναι ο κύριος Μάικλ Γκάλερ. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρησή μου. Έπρεπε να παραστώ σε ψηφοφορία στην άλλη μου επιτροπή. Βρίσκομαι εδώ αρκετό καιρό. Ε, είχα επαφές με την Διακοινοβουλευτική Ένωση ε, στην Ελβετία. Μία από τις εμπειρίες που έζησα ήταν η εξής. Εκπροσωπείται ε, τα κοινοβούλια όλων των χωρών των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι Εκπροσωπείται και χώρες μη δημοκρατικές. Θυμάμαι συζήτηση με τον εκπρόσωπο ε, της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών ε, να οδηγούν αυτοκίνητο. Αυτό τώρα πια ε, έχει ξεπεραστεί, αλλά είναι απλά ένα παράδειγμα. Με όλη την πυρογνωμοσύνη λοιπόν που έχετε, ποιες είναι οι εμπειρίες σας σχετικά με τη συμμετοχή αυτών των μη δημοκρατικών χωρών εσείς προσφέρετε εμπειρογνωσία, σεμινάρια και ε, υποθέτετε ότι ε, όλα αυτά ε, γίνονται σε δημοκρατικό πλαίσιο. Τι γίνεται με την Κίνα. Δεν συμμετέχουν καν, φαντάζομαι, σε συναντήσεις ε, όπου ε, προϋπόθεση θεωρείται το να υπάρχουν επιλογές, το να υπάρχουν θέματα προς συζήτηση. Και αν όχι εκεί, να πιστεύετε ότι ίσως κάποιες μικρότερες ε, αυταρχικές ε, χώρε σε κάποια ολοκληρωτικά καθεστώτα θα μπορέσουν να συμμετάσχουν ε, σε τέτοιε συζητήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Ο κύριος Πίσουλα δεν είναι παρόν. Ε, δίνω το λόγο στην κυρία Χίλτε Βάουτμαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ζήτησα όμως το λόγο. Εγώ θέλω να μιλήσω πάνω στην έκθεση. Ζητώ συγγνώμη, Φιλ. Ωραία, θα πάρω εγώ το λόγο τότε. Ο κύριος Σεμπένιον. Ε, ήμουν εκπρόσωπος ε, στη Διακοινοβουλευτική Ένωση ε, κάποιες φορές. Ε, ε, εκπροσωπώντας την Libre International που ε, έχει ε, καθεστώς ΜΚΟ παρότι είναι ο Διεθνής Οργανισμός Φιλελεύθερων Κομμάτων. Κάποιες από τις παρατηρήσεις μου ήταν ε, παρόμοιες με αυτές του κυρίου Γκάλερ. Αναρωτιέμαι δηλαδή αν υπάρχει η δυνατότητα η Διακοινοβουλευτική Ένωση να προωθεί πιο ενεργά τη δημοκρατία. Συμμετείχα σε μια συνάντηση στο Μπαγκλατές. όπου ε, ακούσαμε ε, να ε, περηφανεύεται η ηγέτη του Παγκλατές ότι θα κάνει μονοκομματικό το κράτος. Η Ζιμπάμπουε και η Βενεζουέλα ε, περηφανεύονταν σχετικά με τις ε, καταπληκτικές επιτυχίες της οικονομίας τους. Ένιωσα όμως ότι υπάρχει και αξία στη Διακοινοβουλευτική Ένωση, μπορεί να συγκεντρώσει ε, ομοειδεάτες πιο πολύ στα περιθώρια παρά στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες να προωθήσουμε τη δημοκρατία. άλλωστε πρόκειται για μια λέσχη κοινοβουλίων, μια ένωση κοινοβουλίων και νομίζω ότι ως τέτοια θα πρέπει να προωθεί ε, περισσότερο την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, έχει επίσης μια πολύ καλή επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα των βουλευτών. Ε, εγώ χρησιμοποιώ την έκθεση, τα συμπεράσματα της επιτροπής αυτής και τα βρίσκω πολύ πολύ χρήσιμα ε, και ε, στον ε, ρόλο μου στην Διεθνή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσατε να έχετε πιο συγκεκριμένο θεματολόγιο. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στον κύριο Ράινχαρτ Μπιουτικόφερ. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, δεν ζήτησα το λόγο. Ε, Διατρέχουμε τώρα τους ε, συντονιστές. Ε, Μαριάννη, παρακαλώ. Τιερή Μαριάννη. Euh, ευχαριστώ. Θα θέσω μία ερώτηση εκ μέρους της ομάδας ε, Ταυτότητα και Δημοκρατία και έχω και μία παρατήρηση. Κυρία μου, σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε στις δυσκολίες και τα προβλήματα πολλών κοινοβουλίων, εθνικών κοινοβουλίων, που εκπροσωπούν όλο και λιγότερο τους τοπικούς πληθυσμούς ή το, ε, τους κατοίκους μιας χώρας. Αναφερθήκατε σε κοινωνικά προβλήματα. Εμείς ανήκουμε στην ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία και έχουμε εκλεγεί στη Γαλλία. Η Γαλλία είναι ένα ιδιάζον παράδειγμα, γιατί ο Εθνικός Συναγερμός ε, με την υποψήφιό του στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών ε, που παρόλο που προηγήθηκε στις περισσότερες ε, εκλογικέ περιφέρειες ε, έχει μόνο 105 βουλευτές στην ε, Εθνοσυνέλευση τη Γαλλική. Και εδώ και ένα χρόνο έχουμε το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων στη Γαλλία που εκφράζει αυτή τη δυσαρέσκεια για την έλλειψη δημοκρατίας στη Γαλλία. Και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ένα μοντέλο δημοκρατικής λειτουργίας που δυστυχώς λάμπει της απουσίας του οπότε θα ήθελα να σχολιάσετε την ε, εσωτερική μας λειτουργία, γιατί αν ε, θέλετε να συνεργαστούμε, φαντάζομαι θέλετε να προωθήσετε ένα δημοκρατικό μοντέλο. Όταν όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένας κανόνας ε, υποτίθεται ότι εφαρμόζεται, όπως είναι ο κανόνας ΔΕΟΝΤ, που διέπει την κατανομή θόκων και αξιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, για τις θέσεις των αντιπροέδρων ή προέδρων επιτροπών και ξαφνικά ως διαμαγείας καταργείται για συγκεκριμένες ομάδες παρόλο που είναι αντιπροσωπευτικές όπως για τη δική μας ομάδα, τη ταυτότητα και δημοκρατία που εκπροσωπούμαστε σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε μάλιστα προηγηθεί σε πολλέ εκλογικέ διαδικασίε, Παρ' όλα αυτά αποκλειόμαστε από αξιώματα εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξαιτία αυτή τη εσωτερική μα λειτουργία. Πώ σχολιάζετε αυτή την κατάσταση, γιατί το να δεσμευτείτε σε μια ασχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να προωθήσετε στον κόσμο τη δημοκρατία ε, και τις σχέσεις με τα εθνικά και διαπεριφερειακά κοινοβούλια, ενώ εμείς οι ίδιοι έχουμε μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν σας φαίνεται κάπως περίεργο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χαβιέρ Λόπες είναι ο επόμενος μου συντονιστής στο κατάλογο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφό μας την κυρία Κουέβας που ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την ευχαριστήσω για το έργο της ε, Διακοινοβουλευτικής Ένωσης ε, ένα φορέα που το θεωρούμε αδελφό φορέα ε, λόγω της πρωτοπορίας στην διακοινοβουλευτική συνεργασία και λόγω της υπερεθνικής λογικής που ασθενιζόμαστε και εμείς ε, με τη συμμετοχή μας σε πολλές πολυμερείς οργανώσεις ε, από το 1945 και μετά. Συμφωνώ με την ανάλυση που κάνατε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η φιλελεύθερη δημοκρατία και για τα φαινόμενα που δυσκολεύουν όλο και περισσότερο την διακυβέρνηση σήμερα. Και θα ήθελα να σας θέσω τρεις ερωτήσεις. Καταρχήν, ως προς την πόλωση που βιώνουμε σε διάφορα κοινοβούλια και εδώ. Ε, μερικές φορές τα εθνικά συστήματα δημιουργούν μια απόλωση με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η δημιουργία συνένεσης, η αναζήτηση κοινών σημείων. Και πραγματικά έχουμε πολλές φορές ε, αφηγήματα μίσους και ανησυχητικά φαινόμενα και στις κοινωνίες. Επίση, η οικουμενική αξία της φιλελεύθερη δημοκρατίας που ήταν αδιάστητη το τελευταίο ε, αιώνα, αλλά δυστυχώ τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει κλονιστεί και φαίνεται ότι έχουμε περισσότερο στρατηγικά τροτά σημεία παρά ε, οικουμενικό χαρακτήρα. Αναφερθήκατε στην τυραννία της αμεσότητας πριν από λίγο. Ε, παλιά είχαμε και τον αυταρχισμό, αλλά έχουμε και πιο σύγχρονες προκλήσεις και σίγουρα η Διακοινοβουλευτική Ένωση είναι διαμεσολαβητής και συνομιλητής ε, και με τα Ηνωμένα Έθνη. Οπότε, τι γίνεται με τα Ηνωμένα Έθνη και την προσπάθεια που κάνουν για την πολυμέρεια χάρη στις ε, ενέργειες και του Γενικού Γραμματέας, τις οποίες εκτιμούμε ιδιαίτερως. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάνκο ζήτησε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Άκουσα με ενδιαφέρον την παρουσίασή σα ιδιαίτερα σε σχέση με τα θέματα τη ισότητα των φίλων και τη εκπροσώπηση των γυναικών στα κοινοβούλια και έχω την εξή ερώτηση σχετικά με αυτό. Κοιτώντα τα μέλη σα τη IPU δηλαδή, πώς έχει η κατανομή στις χώρες εκείνες όπου παρακολουθούμε, παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις και έχετε αρκετά μέλη από τα Αφρικανικά Κοινοβούλια γιατί βλέπω τις εκθέσεις σας ότι στη Ρουάντα έχουμε άνω το 60% εκπροσώπηση γυναικών. Και θα ήθελα να την που σχετικά με τη συμμετοχή των Αφρικανικών Κοινοβουλίων γενικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλατε να απαντήσετε στα ερωτήματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα δημοκρατία. Θα περάσω στα ισπανικά αν μου επιτρέπετε. Ιδιαίτερα μιλώντα για τη δημοκρατία. Έχουμε δύο επιλογές για το πώς θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Η πρώτη είναι η συζήτηση που είχαμε στη Διακοινωνική Ένωση για το κατά πόσον Δημοκρατική χώρα σημαίνει εκλεγμένο κοινοβούλιο. Έθουσες κοινοβουλευτικές, άνω ή κάτω βουλή, όπως ορίζεται υπό την κάθε χώρα. Αλλά γιατί συμπεριλαμβάνουμε χώρες στι οποίε αυτές οι αίθουσες ή αυτές οι βουλές ορίζονται από μια κεντρική αρχή και δεν είναι εκλεγμένες. Στα πλαίσια τη συζήτηση αυτή, εγώ προσπαθώ να έχω μια ρεαλιστική προσέγγιση. Σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως είναι καλύτερο να συμπεριλαμβάνουμε χώρες, να εκπροσωπούνται δηλαδή χώρες μη δημοκρατικές, ώστε να μαθαίνουν τη, τη δημοκρατική πρακτική, παρά να έχουμε μια λέσχη, αν θέλετε, μια ομάδα πιο ομοιογενή και πιο δημοκρατική, αφήνοντα αυτέ τι χώρε απ' έξω, χωρί να μαθαίνουν τη δημοκρατική πρακτική. Κάποιες χώρες διατηρήθηκαν στην Ένωση, εκπροσωπούνται δηλαδή στην Ένωση, που προήλθαν οι κυβερνήσεις τους από πραξικοπήματα. Εάν η ίδια η χώρα δεν ακολουθεί το σύνταγμά της ή τις διατάξεις της, το δίκαιο, το εσωτερικό της, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Από εκεί πέρα, αν δούμε πού οδηγεί αυτή η προσπάθεια, έχει και θετικά αποτελέσματα. Κάποιες από τις χώρες αυτές ξεκινούν, ξεκινούν εξετάζουν μια εκλογική διαδικασία. Το Κατάρ, για παράδειγμα, εδώ και λίγες ημέρες ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει μια διαδικασία εκλογική ώστε να σχηματίσει μια εκλεγμένη βουλή. και στα θέματα της ισότητας των φίλων και των νέων. Είχαμε μια εκστρατεία πριν από λίγα χρόνια, not too young to run, ότι κανείς δεν είναι υπερβολικά νέος ώστε να είναι μέλος του Κοινοβουλίου ή εκλεγμένος. Δεν είναι εύκολες οι προσπάθειες αυτές. Διότι υπάρχει μια τάση προς τον αυταρχισμό, υπάρχει μια λαϊκιστική τάση που τραβάει την προσοχή και γι' αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό χρονικό σημείο η Κοινοβουλευτική Ένωση, τα κοινοβούλια να ανακτήσουν μια εικόνα ενεργούς πρόθεσης, ενεργούς υποστήριξης του κράτου δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δημοκρατικού πλαισίου, της δημοκρατικής κοινωνίας. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλους μας. Και πρέπει επίσης να κάνουμε μια προσπάθεια προς μια άλλη κατεύθυνση. Όχι να μαθαίνουμε τόσο σε χώρες που δεν είναι δημοκρατικές πώς να είναι, αλλά να ανακτήσουν τη δημοκρατικότητά τους χώρες που υπήρξαν πάρα πολύ δημοκρατικές και που σήμερα έχουν υποχωρήσει έναντι πιο αυταρχικών συστημάτων. Πρέπει λοιπόν να διαφοροποιήσουμε την προσέγγιση μας ανάλογα με τους συνομιλητές που έχουμε απέναντί μας. Κι άλλο ένα θέμα στην Ένωση είναι η Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Κοινοβουλίων. Μερικές φορές σκέφτεται κανείς ότι το να είναι βουλευτής είναι κάτι το... Ε, έχει μια έγκλη. αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να μάχεται ο κάθε βουλευτής, το κάθε μέλος του Κοινοβουλίου, ώστε να ερευνά, να εξετάζει κατά πόσον προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών αλλά και των μελών του Κοινοβουλίου. Στον 21ο αιώνα που βρισκόμαστε έχουμε άνω των 600 καταγγελιών παραβιάσεων των δημοκρατικών δικαιωμάτων μελών του Κοινοβουλίου. Ελευθερία έκφραση, αλλά και πολύ σοβαρών περιπτώσεων ακόμα και κράτησης και δολοφονία μελών των κοινοβουλίων. Και στην Επιτροπή αυτή θα μπορούσαμε να έχουμε ένα διάλογο προσκαλώντας κάποια από τα μέλη της Επιτροπής εκείνης της δικής μας, ε, ε, ώστε να σας εξηγήσουμε τη δουλειά, την προσπάθεια που κάνουμε. Γιατί μερικές φορές πραγματικά είναι η διαφορά ανάμεσα στην επιβίωση και στο θάνατο για κάποιους από τους συναδέλφους μας. Νομίζω ότι η Διακοινοβουλευτική Ένωση έχει τεράστιες δυνατότητε και μερικές φορές ούτε εμείς οι ίδιοι δεν τις αντιλαμβανόμαστε και σας δίνω ένα παράδειγμα. Τι θα συνέβαινε αν μία μέρα οι 46.000 βουλευτές στον κόσμο αποφάσισαν να συνεργαστούν με κοινό πρόγραμμα, με κοινή στρατηγική προς μια κοινή κατεύθυνση. Νομίζω ότι πραγματικά θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό παράδειγμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ε, ελπίζω να μπορέσουμε κάποια στιγμή να έχουμε τόσο αποτελεσματική συνεργασία στην Ένωση. Αν έχουμε δημοκρατικό έλλειμμα, με ρωτάτε, ναι έχουμε. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και να το αναγνωρίζουμε. Έχουμε υποχώρηση έναντι της δημαγωγίας και του λαϊκισμού. Αλλά πρέπει να είμαστε και αυτοκριτικοί, πρέπει να είμαστε ειλικρινεί σχετικά με το πώς υποχωρούν οι θεσμοί μας, τα θεσμικά μας όργανα που δεν είναι απόλυτα προσβάσιμα για τις γυναίκες και για τους νέους. Ενώ πολύ συχνά βλέπουμε ότι η πρόσβαση των μη όμικρων σε κάποιες χώρες είναι αρκετά εξασφαλισμένη, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι πολλά κοινοβουλία δεν έχουν καθόλου καλή άποψη για αυτές, για τις μη όμικρων. Η ελευθερία της έκφρασης είναι κάτι που δεν μπορεί να το ξεχωρίσει κανείς από τη δημοκρατία. Ακούμε όμως συζητήσεις και αφηγήματα που έχουν απήχηση τελικά στην κοινή γνώμη και ε, δημοκρατία δεν είναι απλώς το να προσέρχονται οι πολίτες στις κάλπες. Αλλά έχει να κάνει με τη συμμετοχή, με τη συμπερίληψη. Όχι μόνο στο θεματολόγιο της ανάπτυξης για το 2030. Όχι μόνο απέναντι σε προβλήματα που είναι πολύ επίγοντα παγκοσμίω. Όχι μόνο για τα θέματα των γυναικών και των νέων, αλλά πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε τις διαδικασίες λήψης απόφασης για την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχικότητα για όλους. Να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ των εκπροσώπων και των πολιτών, του κόσμου και των βουλευτών. Το Κοινοβούλιο στην Κύπρο, για παράδειγμα, έχει μια πρωτοβουλία για το παράλληλο κοινοβούλιο. Με θεματικές που αφορούν στην κοινωνία, με ομάδες, αν θέλετε, συζήτησης, που, που καταλήγουν σε προτάσεις, σε πρωτοβουλίε οι οποίες υποβάλλονται προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο. Τον Καναδά επανεξετάζουν την μέθοδο με την οποία ορίζονται τα μέλη της Άνω Βουλής, ώστε οι πολίτες να μπορούν να συμμετέχουν πολύ πιο ενεργά και ανοιχτά, χωρίς αυτό να επηρεάζεται από τα πολιτικά κόμματα, παρά μόνο από την ικανότητα των πολιτών. Πρέπει να, είμαστε, να εξασφαλίζουμε ότι η δημοκρατία μας θα είναι αποτελεσματική. Όχι ναι ή όχι δημοκρατία, αλλά δημοκρατία πώς. Πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική η δημοκρατία για να είναι αποτελεσματική. Η, Διακοινοβουλευτική Ένωση είναι ο, θεσμός, ε, ο πολυμερής θεσμός ο αρχαιότερος, αλλά ως τέτοιος πρέπει και να εξυγχρονίζεται. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και επιμένω σε αυτό. Μιλούμε για πόλωση παγκοσμίω, είναι αλήθεια. Γι' αυτό ισχύει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Και σε μερικές χώρες ε, δεν υπάρχει τόσο έντονη η λαϊκή εκπροσώπηση και είναι εύκολο να το εξηγήσουμε το θέμα της πόλωσης. Και στην δική μου περιοχή, στη Χιλή, ουσιαστικά δεν έχουμε διαφθορά και τα ελάχιστα κρούσματα διαφθοράς ε, πατάσσονται και τιμωρούνται. Η μεσαία τάξη είναι εύρωστη και κεντροαριστερά κόμματα με πολύ ενδιαφέρον κοινωνικό πρόγραμμα διακυβέρνησαν για πολύ καιρό. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κοινωνική διαμαρτυρία που ζητά ουσιαστική άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό και με ενδιαφέρει ο διάλογος με τους χιλιανούς ε, βουλευτές. Γιατί τα πολιτικά κόμματα κατέληξαν όλα στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει σήμερα να διαρωτηθούμε πού κάναμε το λάθος και πώς θα διορθώσουμε την κατάσταση. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό που μας λείπει είναι να αντιληφθούμε ότι αυτή η πόλωση δεν είναι εξορισμού κακή. Αν αντιληφθούμε ότι η φύση ενός κοινοβουλίου έγκυται στο διάλογο και στην ανταλλαγή απόψεων. Ο κόσμος μερικές φορές μας επικρίνει, γιατί λένε εσείς ε, ξοδεύετε όλο σας το χρόνο με τη συζήτηση. Αλλά η συζήτηση είναι μέθοδος εργασία σε ένα κοινοβούλιο και θα πρέπει να μας οδηγήσει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Και γι' αυτό ψηφίζουμε, γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαδικασία και γι' αυτό ψηφίζουμε. Και η μέθοδος η δημοκρατική είναι η καλύτερη. Εμένα δεν με φοβίζει ούτε η αντιπαράθεση ούτε η πόλωση. Αυτό που με προβληματίζει και με ανησυχεί είναι ότι σήμερα το πολιτικό αφήγημα δεν είναι η συμφωνία και η κοινοβουλευτική συζήτηση, αλλά η υποδάβληση ε, διαμάχης και η μεταφορά της στους δρόμους. Γιατί με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε κάποιες ε, εθνοκαθάρσεις και τις ε, σοβαρότερες ε, τραγωδίες της ανθρωπότητας. Με προβληματίζει και με ανησυχεί αυτό που συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με αυτό το αφήγημα του μίσους. Και κάτι τέτοιο βιώνουμε και στα βόρεια σύνορα της χώρας μας, γιατί όποιος παίζει με το μίσος θα το βρει μπροστά του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση και την, ε, τις ε, διαπραγματεύσεις και τις επαφές με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τα Ηνωμένα Έθνη και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είμαστε υπέρ τη πολυμέρεια. Δεν είναι εύκολο. Προσκρούμε στην αντίθεση και στην αντίσταση μερικών κυβερνήσεων. Που σίγουρα αυτό το θέμα δεν του είναι ιδιαίτερα προσφυλέ. Αλλά θα πρέπει να βρούμε κάποιο κάποια σημεία συνεργασίας. Εμείς έχουμε κάθε Φεβρουάριο ε, τέτοιες συζητήσεις. Ε, επίσης έχουμε το, το Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου και την, Εθνική Συνέ... την ε, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έχουμε μια εβδομάδα για την κατάσταση των γυναικών. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις πρωτοβουλίας ε, και συνδιοργάνωσης με τα Ηνωμένα Έθνη που είναι πολύ χρήσιμες ευκαιρίες ανταλλαγής απόψεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επισκεφτήκατε και που μοιραστήκατε μαζί μας ε, τις απόψεις σας σχετικά με την κατάσταση της δημοκρατίας. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας ξαναφιλοξενήσουμε εδώ για να συνεχίσουμε τη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στις διάφορες χώρες ε, και τη συνεργασία μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης ε, και θα δώσω αμέσως το λόγο στον David McAllister.